με βάση το άρθρο 74 του κανονισμού ε, μαζί ε, υπέγραψα ε, τέσσερις νομικές πράξεις οι οποίες έχουν εγκριθεί. Οι τίτλοι των νομικών πράξεων θα δημοσιευθούν στα πρακτικά της συνεδρίασης αυτής. Και τώρα περνάμε στο πρόγραμμα εργασιών μας με βάση το άρθρο 137 στις